Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Πρώτον, το τέσσερα, Για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη. Οι τροπολογίες υποβλήθηκαν έγκαιρα και η έκθεση λοιπόν επίσης υποβλήθηκε έγκαιρα. Επειδή σήμερα έχουμε πολλές ψηφοφορίες και ορισμένες πολύ περίπλοκες, πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, θα ήθελα να ελέγξουμε τις ηλεκτρονικές κάρτες και την παρουσία. Οπότε σας παρακαλώ πρώτα να κάνουμε ένα τεστ. Παρακαλώ ε, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Λοιπόν, είμαστε 41 βουλευτές, 41 βουλευτές, βουλευτές παρόντες. Αυτός είναι ο αριθμός των μελών που πρέπει να έχουμε. Όλοι έχετε τις κάρτες σας. Οπότε, είμαστε έτοιμοι. Πρώτον, τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ Κατά. Συγγνώμη. Τροπολογία 16. απόχέ, Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. το τελευταίο τμήμα της τροπολογίας 20 μπορεί να ε, ψηφιστεί ως συμπλήρωση. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και το τελευταίο τμήμα της 23 θα μπορούσε να θεωρηθεί προσθήκη στο κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 55 υπέρ με συγχωρείτε α καταπίπτει οπότε είμαστε στις 50, στην 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα να ψηφίσουμε το τροποποιηθέν κείμενο ηλεκτρονικά άρχεται Ε, πέρας. Α, λειτουργεί το μηχάνημά σας. Α, ωραία. Οπότε, σας παρακαλώ, άρχεται εκ νέου ψηφοφορία. Πέρας.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 Πέρας. Ωραία. Ωραία ήταν σαφής ε, νομίζω η κατάσταση. Συμβαστική για τον μπλοκ 2 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική για τον μπλοκ 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Α, καταπίπτει. Και 48. Οπότε περνάμε στην 51. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε Αιτιολογικές σκέψεις και συγκεκριμένα τροπολογία 12. Υπέρ παρακαλώ. Συγγνώμη τι είπατε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Υπάρχει μία ε, προφορική τροπολογία την οποία ε, δεν είδα είναι τροπολογήση, τροπολόγηση του άρθρου 5, είναι η προφορική τροπολογία 1. Έχει κανείς αντίρρηση να συζητηθεί. Ωραία, να την ψηφίσουμε τότε. Ποιοι είναι υπέρ της, ε, της προφορικής τροπολογία 1, παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στις ιδεολογικές σκέψεις. Πρώτα απ' όλα τροπολογία 12. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην προφορική τροπολογία 4. Υπάρχουν αντιρρήσεις να ψηφιστεί. Όχι. Ωραία να ψηφίσουμε ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 2 έχει αντίρρηση κανείς να ψηφιστεί όχι ωραία ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε τώρα την τροποποιηθής γνωμοδότηση άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. 34 υπέρ. Ε, ευχα... Ε, συγχαρητήρια και πάλι στην εισηγήτρια. Οπότε τώρα περνάμε στην ψηφοφορία για το σημείο 6 εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής ε, στις πρωτοβουλίες δημοσίου ιδιωτικού χαρακτήρα. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Είναι συμβιβαστική τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40, 58 συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 58. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην ΙΜΚΟ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά α, κατά Μάλιστα, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία ΙΜΚΟ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία ντεβε 11 υπέρ α με συγχωρείτε με συγχωρείτε καταπίπτει εφόσον ενεκρίθη συμβαστική 3 συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Και τώρα 70 υπέρ. κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται τροπολογία 78 α καλά καλά να ελέγξουμε την 77 άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 5 ως προσθήκη υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 4 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ας ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της ΣΥΜΚΟ 4 άρχεται Πέρασε. εγκρίνεται Ντεβε 7. Α, καταπίπτει. Συμβαστική 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική Επτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΔΕΒΕ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΔΕΒΕ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 97 υπέρ κατά Ας την ελέγξουμε γιατί δεν σηκώνετε όλα τα χέρια σας. Ελέγχουμε την 97 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 22 ψήφους υπέρ. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 15 ως προσθήκη υπέρ. Κατά Λοιπόν, λοιπόν, σας παρακαλώ και πάλι. Υπέρ ΙΜΚΟ 15. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. 10, 10 βεβαίως. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε... Τροπολογία 110 υπέρ. Κατά. Λοιπόν, παρακαλώ, 110 ε, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ντέβε 14. Υπέρ. Συγγνώμη. Α, συγγνώμη. Καταπίπτει γιατί έχει εγκριθεί η συμβαστική 10. Ωραία. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 117 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Για την 117. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 118 υπέρ. Κατά. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε. Θέλω να είμαι σαφέστατος. 118. Διαχειρός. Παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 121. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογικές σκέψεις τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά Αποχές. Έλεγχος. Τροπολογία 24. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 1. Υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τριάντα ένα υπέρ Όχι, δεν εγκρίθηκε 29. 31 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ήμκο 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά, κατά αποχές 34 τροπολογία με προφορική τροποποίηση δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ποιοι είναι υπέρ λοιπόν κατά αποχές εγκρίθηκε ΙΜΚΟ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 38 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 44 υπέρ κατά Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 44 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε ντεβε μπλοκ 2 3 4 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν ντεβε μπλοκ 6 9 και 10 υπέρ αυτών κατά θα ελέγξουμε λοιπόν ψηφίζουμε 6, 9, 10 ντεβε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκαν ντεβε μπλοκ 12 και 13 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. και με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε θερμά συγχαρητήρια εισηγητά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 Περνάμε τώρα και θα ψηφίσουμε την έκθεση ενδιάμεσος απολογισμός TTIP. Γιάννικ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν θα μακρηγορήσω για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα, μόλον ότι είχαμε προθεσμία χθε μέχρι τις 12 το μεσημέρι για την κατάθεση τροπολογιών και συμβαστικών τροπολογιών. Ορισμένε πολιτικέ ομάδε υπερέβησαν αυτή τη χρονική προθεσμία, συγκεκριμένα μια συμβαστική πρόταση από τον ίδιο τον πρόεδρο. Θα ήθελα όμω να μιλήσω λίγο περισσότερο για την το πώς ακολουθείται η σειρά στις τροπολογίες, ιδίω όσον αφορά την τροπολογία 50, την συμβαστική τροπολογία 50 που αναφέρεται στο ISDS. Νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρους κανόνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες εκείνες οι οποίες απέχουν περισσότερο από το αρχικό κείμενο και που έχει καταθέσει ο συγητής. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε μια εντελώ διαφορετική παράλογη κατάσταση, όπου τελικά βλέπουμε ότι ο κατάλογος ψηφοφορίας και η σειρά μάλλον των τροπολογιών για τις διάφορες συμβαστικές τροπολογίες όσον αφορά το 50 στην πράξη έχει οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο προκειμένου να διευθετήσει περισσότερο τη σημερινή ψηφοφορία και όχι τους κανόνες. Επομένως, η συμβαστική τροπολογία 50 από το EFTD, την ΚΟΕ e και τους πράσινους θα πρέπει, όπως λένε οι κανόνες, να ψηφιστεί πρώτη. Ευχαριστώ. Ähm, äh, Ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, Τζανίκ πρέπει να πω ότι σαφώς οι κανόνες τα άρθρα νομίζω είναι το 170 άρθρο του κανονισμού που λέει ότι οι τροπολογίες που απέχουν περισσότερο από το αρχικό κείμενο εκείνες πρώτα θα πρέπει να ψηφιστούν καταρχήν και θα θυμάσαι σίγουρα στο αρχικό μου κείμενο γίνεται λόγος για το ότι το ISDS ε, δεν είναι αναγκαίο για την TTIP και έτσι πολύ όμοια με την τροπολογία της ΓΚΟΕ και των Πρασίνων ε, εμπίπτει στο πλαίσιο αυτό και έτσι πριν από το αρχικό κείμενο θα πρέπει λόγω της παρέκκλησης να ψηφιστούν. Εσύ έχεις τον λόγο. Συνεπώς το προτινόμενο κείμενο από τον πρόεδρο, τον εισηγητή, είναι το κείμενο το οποίο απέχει περισσότερο τελικά από το αρχικό κείμενο το οποίο υπέβαλε ο ίδιος ο εισηγητής στην αρχή διαπραγματεύσεων. Επομένως το αίτημά μας είναι το ακόλουθο. Η πρώτη συμβαστική η οποία προτείνεται να έχει ονομαστική ψηφοφορία, να γίνει μονομαστική κλίση. Δηλαδή για το 50α να έχουμε ονομαστική κλίση. Ευχαριστώ. Le délai est aussi dépassé depuis longtemps, chers collègues. Μα αγαπητέ συνάδελφοι, έχουμε περάσει και την προθεσμία κατάθεση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Helmut. Helmut, παρακαλώ. Ja, selbst, also wenn Ναι, ακόμα και αν έχει λήξει έστω η προθεσμία όπως ακούστηκε μόλις θα πρέπει να εμείνω και να επιμείνω ότι roll call vote η, ονομαστική κλίση μια και ε, ε, το βράδυ κατατέθηκε ο συμβιβασμός και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε θα πρέπει έτσι να αντιμετωπίσουμε πριν από τις 12 κατατέθηκε μετά όμω από την κατάρτιση του πίνακα ψηφοφορίας μετά από την ολοκλήρωση του πίνακα ψηφοφορία που διανεμήθηκε όμως για αυτά τα πράγματα έχουμε σαφείς κανόνες και αυτοί θα εφαρμοστούν εδώ τώρα. Αυτοί θα ισχύουν. Όταν μια ονομαστική, διανομαστική κλίσης ψηφοφορία ζητείτε, τότε πρέπει ένα τέταρτο των μελών να εγκρίνουν το αίτημα και θα το ελέγξουμε αυτό αν πράγματι συμβαίνει. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν. Είναι 11 σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Ποιοι είναι υπέρ της ονομαστικής κλίσης για το 50α. Παρακαλώ όσοι είναι υπέρ να το αναφέρουν. Εσείς πιο πριν παρακαλώ. Ήθελα απλώ να επιβεβαιώσω ότι ο τελικός κατάλογος ψηφοφορίας δόθηκε στις 12.48 χθε τα ξημερώματα ή ενδεχομένω πήγαινε καλά το ρολόι του Κοινοβουλίου. Πάντως όλοι λάβαμε στις 12.48 τα μεσάνυχτα το τελικό κατάλογο ψηφοφορίας. Ακούστε, ε, πρόκειται για το θέμα της κατάθεσης των τροπολογιών ως προθεσμία, 12 ήταν η προθεσμία. Δυστυχώς η κατάρτιση του πίνακα ψηφοφορίας χρονοβόρησε και είχα και εγώ και την ευχαρίστηση μέχρι τη μία να είμαι στο Κοινοβούλιο ώστε να μπορέσω να διοργανώσω αυτά τα ζητήματα, να τα διευθετήσω και λόγω των διαπραγματεύσεων και των διεργασιών δημιουργήθηκε μια έκτακτη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει και πάλι τώρα για αυτή την τροπολογία ονομαστική ε, ψηφοφορία για το 50α. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν να γίνει ονομαστικά η ψηφοφορία. Δέκα. Δέκα που καταμετρήθηκαν και είδαμε και καταμετρήσαμε. Δεν ε, υλοποιείται ο όρος της απαρτίας λοιπόν. Μπορούμε να το ελέγξουμε αν θέλετε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για να διαπιστώσουμε πόσοι είναι υπέρ. Πέρας ψηφοφορίας. 11 ε, είναι, μάλιστα. Ε, κατά τούτο λοιπόν τώρα κάποιος άλλαξε άποψη, άλλαξε γνώμη και εντάξει θα έχουμε λοιπόν με ονομαστική ψηφοφορία τη διεξαγωγή. Εντάξει, προχωράμε. Να υπενθυμίσω και κάτι άλλο τώρα πρώτα. Προσπάθησα με ένα πνεύμα ένταξης όλων των αιτήματων να αντιμετωπίσω τα αιτήματα. Είχαμε έξι με τους σκιώδεις εισηγητές διαπραγματεύσεων, τρεις γύρους ε, με την εισηγήτρια, με τις εισηγήτρες, εισηγητές ε, των κοινοβουλευτικών επιτροπών που συνέταξαν γνωμοδοτήσεις, 13 εν συνόλο. Μεγάλη λοιπόν εικόνα, ολοκληρωμένη εικόνα με απόψεις που εντάχθηκαν στην διαδικασία συζητήσεων και διαβουλεύσεων με τις πιο διαφορετικές απόψεις για την TTIP. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το δυνατόν πιο ενωμένοι θα πρέπει να τοποθετηθούμε ως Ευρωκοινοβούλιο και έτσι το δυνατόν τις περισσότερες ε, γνώμες και τοποθετήσεις των συναδέλφων να τις συμπεριλάβουμε ώστε να δώσουμε ένα σαφέστατο μήνυμα έναντι των εταίρων και διαπραγματευτών από την άλλη όχθη, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού να περάσει ένα σαφέστατο μήνυμα. Κατά τούτο ήταν λοιπόν μια σε βάθος εντατική αλλά και διαφανέστατη διαδικασία που καταλήγει σήμερα στην ψήφιση, στην ψηφοφορία. Έχουμε τα τμήματα πινάκων ψηφοφορίας. Θα τεθούν σε ψήφιση όλα αυτά τα θέματα των επτά πινάκων και όσοι ήθιστε με τις παραγράφους, τα εδάφια και ξεκινάμε πρώτα πρώτα ψηφίζοντας με τη συμβαστική τροπολογία 13 λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ της συμβαστικής 13. Παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε η συμβαστική 13. Περνάμε στη συνέχεια στην τροπολογία 252 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 253 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 254 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό 14 υπέρ Παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Ωραία. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 268. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 270. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε στο συμβιβασμό 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην 278 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε στη συμβιβαστική τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στη συμβαστική τροπολογία 16 α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε τώρα στην τροπολογία 289 υπέρ είναι γλωσσική η διατύπωση είναι που ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 291 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε. Εντάξει, ψηφίζουμε την 291. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας συγγνώμη, ε, έχουμε, ε, ξεπερνάμε τις ψήφους μας. 42, ε. Α, εντάξει, ωραία, εντάξει, είμαστε στο όριο. Απορρίφθηκε. 294 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 298 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε και 300 τροπολογία 300 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε και έτσι περνάμε τώρα στον πίνακα ψηφοφορίας υπαριθμών 2 301 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβασμός 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στην τροπολογία 312 συγγνώμη 310 πρώτα 310 λοιπόν υπέρ κατά έλεγχος ωραία ψηφίζουμε την 310 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε τροπολογία 312 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε περνάμε στην τροπολογία 315 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε στη συνέχεια θα περάσουμε στην τροπολογία 325 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 329 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 330 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 332 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 338 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 345 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 346 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 347 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 351 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ Κατά. Θα ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και έτσι καταπίπτει η 20α συμβαστική τροπολογία. Και περνάμε στον συμβιβασμό 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 381 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 384 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 386 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Και περνάμε τώρα στον συμβιβασμό 23α. Υπέρ, κατά, κατά παρακαλώ. Εσείς όχι. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Κατά. Μία ψήφος εναντίον. Εντάξει. Ωραία. Αποχές με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε. 23α. Πολύ ωραία. Και περνάμε τώρα στην 421 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 423 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 424 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 425 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 426 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβαστική τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική τροπολογία 24α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 437 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 440 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 441 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 442 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Συμβαστική τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τε, τροπολογία 455 η λίμπε 1 βιτ αλφα. υπέρ, υπέρ αυτών κατά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 455 και 1 αλφα λίμπε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκαν. 456 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κα, δεύτερο, κατά, συγγνώμη, κατά αποχές θα ελέγξουμε πρώτο τμήμα ψηφίζουμε τις 456 άρχεται πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα δεύτερο τμήμα τώρα τις 456 καταπίπτει αυτό εντάξει τροπολογία συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε στην 466 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβαστική τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές ομόφωνα εγκρίθηκε εξαιρετικά. Πολύ ωραία. 482 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 483 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 485 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε άφετ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 510. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τώρα 510 είχαμε πει. Εντάξει να ελέγξουμε. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 510 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε μάλιστα. Εντάξει. Ε, αυτό που βλέπω λέω. Και το είδα σωστά. 512 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 514 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Εντάξει, τώρα πάμε στη συμβαστική τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και πάμε στην 528 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε. 528 τροπολογία δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και τώρα 536 και αυτή σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και τώρα ο πίνακας ψηφοφορίας 3 Καταρχήν 539 υπέρ. Τροπολογία 539. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 540 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 562 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 563 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 564 υπέρ κατά σαφές το αποτέλεσμα θα έλεγα εγκρίθηκε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 564 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 566 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 5 Συγγνώμη, 569. Η 569 είναι μια προσθήκη, ως προσθήκη μπορεί να ψηφιστεί. Ποιοι είναι υπέρ της 569. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Και τώρα πάμε στην 567. 576 ε, με συγχωρείτε υπέρ κατά απορρίφθηκε πάμε στην 580 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 581 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 583 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 584 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 585 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 586 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 587 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Και πάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 599 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 600 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 601 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 609 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε μάλιστα πολύ καλά εντάξει ωραία ωραία τώρα 617 παρόμοια με την ΛΥΜΠΕΕΝΑ θα έρθουμε ύστερα σε αυτήν. Ποιοι είναι υπέρ τη 617. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 618 υπέρ. Κατά. απόχέ Απορρίφθηκε. Και περνάμε στον πίνακα 4. Ψηφοφορία 4. 620 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 621 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 628 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 629 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Αλλά ας ελέγξουμε. Την 6.29. Άρχεται. Πέρας. Α, παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Συμβαστική 38α. Ε, θέλουν να πούν τίποτα αυτοί που την, προτε... την προτείνανε. Όχι γιατί θεωρώ ότι κάτι θα θέλατε να πείτε. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Εδώ βλέπω είναι ELK ECR, ALDE. Στο κατάλογο μας είναι σωστό αυτό που έχω εδώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Έχει αποσυρθεί από τον 38α το ELK Συγγνώμη, συγγνώμη αν δεν το μάθατε, αλλά το, ε, σας ενημερώσαμε κανονικά. Ωραία, 38α. Είναι μόνο από το, από, τους, από το ECR και την ALDE. Μαρίκη, γιατί κουνάς το κεφάλι σου. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι αυτό το τμήμα της γενικότερης σύγχυσης. Μπορούμε να ψηφίσουμε πάντως τροπολογία αυτή. Πάντως, η ισορροπία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τέλο πάντων την 38. Εγώ την έχω αποσύρει και από το δικό μου τον κατάλογο βέβαια. Δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Πρέπει να την ψηφίσουμε ή όχι. Πρόεδρος, ωραία να την ψηφίσουμε. Υπέρ. 38α, έτσι, αυτή ψηφίζουμε. 38α. Ε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα, σημαστική 38 υπέρ κατά αποχές. Ε, στην την ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 38. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε τώρα, 6.42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6.44 καταπίπτει, οπότε συμβαστική 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται οπότε 6.57 υπέρ α παρακαλώ Μαρίτια να ζητήσω ένα τεχνικό έλεγχο σε αυτό το σημείο, γιατί η τροπολογία 6 για το 144 θα κατέπιπτε αν η 42 είχε εγκριθεί, αλλά απορρίφθηκε εξ αρχής νομίζω αυτή, άρα πρέπει να την ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι. 644. Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Απορρίφθηκε 642, άρα πρέπει να ψηφίσουμε την 644. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 643 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε ωραία ελέγχουμε την 6.45 άρχεται α την 6.43 ήθελες καλά εντάξει γιατί όχι αυτή τη δουλειά κάνουμε 6.43 την 6.43 ελέγχουμε άρχεται Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα να ελέγξουμε την 6.45. 6.45. Άρχεται. Πέρας. Mm, mm. Απορρίπτεται. 6.46. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 40 λοιπόν. Υπέρ. Α, την ψηφίσαμε. Ναι, την ψηφίσαμε. Καλά. Εντάξει τώρα, εντάξει. Επειδή άλλαξε η σειρά. Να είμαστε λοιπόν απόλυτα τυπικοί. Ε, 40 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 6.57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτω. Συμβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 665 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 η οποία έχει συνδυαστεί με την αρχική 42β. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην 677 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η επόμενη καταπίπτει. Συμβαστική 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην 693 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 678 καταπίπτει 694 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 700 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 701 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έξι η 695 μπορεί να θεωρηθεί προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 708 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 708. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7-16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 717 7-17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 718 7-18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 729 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 730 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 748 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 50α. Έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Μάλιστα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 ψήφοι υπέρ. Οπότε καταπίπτουν πάρα πολλέ. Περνάμε στην συμβαστική 51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην 807 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 808 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 810 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Την 810. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 811 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 813 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 51β. 51β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα... Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Πέρασα μία. Με συγχωρείτε, αλλά έχουμε δύο διαφορετικούς καταλόγους. Να συντονιστούμε. Γιατί εγώ δεν έχω μια τροπολογία εδώ. Και δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό γιατί είναι και από πλευρά σοσιαλιστών μάλιστα. Η 803. 803 πρέπει να ψηφιστεί. Ναι, ναι, ναι, αλλά κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορετικές ε, εκδοχές του κειμένου. Ας ψηφίσουμε την 803. Ποιος είναι υπέρ της 803. κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα έχουμε μια που δεν την είδαμε μας ξέφυγε είναι 814 του κυρίου Προύστ υπέρ 814 814 κατά αποχές απορρίπτεται οπότε Οπότε, απότε τώρα όμως, έχουμε και την 816. Υπέρ παρακαλώ. Ωραία, ωραία. Ο κύριος Προύστ θέλει να ελέγξουμε την 814. Άρχεται για την 814. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε την 816. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε, όπως γνωρίζετε, στο τμήμα 5. Έχουμε την τροπολογία 823. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ομόφωνα. Οπότε έχουμε την 845 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 846 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 848 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 847 υπέρ 847 υπέρ παρακαλώ κατά να ελέγξουμε ελέγχουμε την 847 άρχεται πέρας απορρίπτεται 851 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 54 υπέρ κατά κατά παρακαλώ ωραία ωραία και αποχές ωραία εγκρίνεται με λίγες αποχές και τώρα Συμβαστική 55. 55 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οκτώ 63. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 871 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 875 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 876 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 877 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 878 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 879 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, έχει προταθεί να ψηφιστούν ε, από κοινού οι άλλες όλες οι άλλες α δεν συμφωνεί δεν συμφωνεί ε, η συντάκτρια ωραία 882 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 883 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 884 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 885 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 886 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 887 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 888 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 889 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 890 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 891 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 892 υπέρ Κατά αποχέ απορρίπτεται. 8-9-3 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 8-9-4 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 8-9-5 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 8-9-6 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται 897 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 898 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Και περνάμε τώρα στον πίνακα ψηφοφορίας 6 αγαπητοί συνάδελφοι γνωμοδοτήσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών που όπως είπαμε στην αρχή αρχή η ένταξη ήταν ε, ολοκληρωμένη να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα και συμβαστικές τροπολογίες. Ψηφίσαμε συμβαστικές τροπολογίες και κατά τούτο καταπίπτουν πολλά σημεία. Σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες ρητά γίνεται αναφορά το ότι υπάρχουν επιμέρους συμπληρώσεις που πρέπει να ψηφιστούν. Γι' αυτό έχουμε αυτό τον πίνακα ψηφοφορίας τώρα και έτσι θα κάνουμε το, έτσι θα προχωρήσουμε. Από την ΑΦΕΤ έχουμε πρώτα το πρώτο τμήμα του άρθρου 1 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα καταπίπτει ναι καταπίπτει έτσι διότι η συμβιβαστική τροπολογία 13 είχε εγκριθεί. ΔΕΒΕΠΕΝΤΕ ΔΕΒΕ5 λοιπόν ξεπερνά το, την εμβέλεια, γι' αυτό προτείνω να απορριφθεί, αλλά ψηφίσουμε. Ποιοι είναι πρώτα, παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίφθηκε η ΔΕΒΕ5. Περνάμε τώρα στην έκον ε ή το είχαμε συζητήσει και στις διαβουλεύσεις μας ως προσθήκη στο 24α στην 24α θα θεωρείτε ποιοι είναι υπέρ κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά έκον ή ψηφίζουμε Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε το ΕΚΟΝ ή e, το I. So, dann kommen wir zu Empel 3. Auch dort müssen wir einzeln abstimmen, wer es darf. Επιτροπή Απασχόλησης 3. Και εδώ πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίφθηκε το Empel 3. Ωραία. Περνάμε τώρα στο τελευταίο τμήμα Εμπλ 6 τελευταίο τμήμα που επιμέρους ψηφίζουμε ξεχωριστά ως προσθήκη στην μόλις εγκριθήσα τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 38. Ποιοι είναι υπέρ του ΕΜΠΛ 6. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά ψηφίσουμε ηλεκτρονικά να δούμε τι απογίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. ΕΜΠΛ 6 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Η ισοψηφία απορρίφθηκε. Και περνάμε στην ΕΜΠΛ 7 σύσταση υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Προχωράμε και φτάνουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ΕΝΒΙ. Λοιπόν, ΕΝΒΙ 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 2, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 3, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 4, υπέρ, και πάλι υπέρ 4, NV4 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. NV5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. NV6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. NV7 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. NV8 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε Act NV8 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Τέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε το NV8. Περνάμε NV9 υπέρ. Κατά Και αυτό θα το ελέγξουμε. NV9. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Και περνάμε στην NV10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. NV11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Ένβη, αιτιολογική σκέψη Β, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Ένβη, το C, recital C, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ένβη, recital E, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. F, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. H, υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε I υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε J υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε K υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε NVL ε. υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε NVO υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε NVP υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Q υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε αιτιολογική σκέψη R υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε S υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε T υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε U υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Β υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε W υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε X υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Y υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Z υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. α υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. AB υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. AC υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. AD υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AE ε, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AF ε, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε G ε, υπέρ κατά κανείς εναντίον AG υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AH υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AI AI υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AJ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AK υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AL υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AM υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AN υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε NV1 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε λοιπόν NV4 και υπενθυμίζω είχαμε τη συζήτηση που είχε διεξαχθεί αν αυτό προσθήκη θα ενταχθεί στην τροπολογία 32 ή όχι και κατά τούτο λοιπόν εδώ τίθεται η δυνατότητα να έχουμε σε τμήματα ψήφιση. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν της NV4. Ποιοι είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Να ελέγξουμε. Πολύ καλά. Δεύτερο τμήμα NV4. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Λοιπόν, το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και με το NV5, τροπολογία NV5, δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος, NV5, κατά αποχές, εγκρίθηκε. NV7, προσθήκη, συμβιβαστική τροπολογία 33 είναι υπέρ αυτού του τμήματος, δευτέρου τμήματος του NV, της NV7 τροπολογίας. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. NV7 δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Λέει ο Αλμπέρτο και έτσι γίνεται και λοιπόν απορρίφθηκε. Ένβη 8 τροπολογία ως προσθήκη στη συμβαστική τροπολογία 22. Ποιοι είναι υπέρ της Ένβη 8. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Ένβη 10 ως προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ της NV10 κατά αποχές απορρίφθηκε περνάμε στην ένβη 13 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την ένβη 13 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ήτρε. Ήτρε 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ήτρε 3. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Περνάμε στην Ήτρε 6. Μπορεί ως προσθήκη να ενταχθεί στην συμβαστική τροπολογία. Πείτε εσείς. Λυπάμαι. Λέει εδώ ότι θα ψηφίσουμε λέει ξεχωριστά. Ποιο τμήμα θα ψηφίσουμε ξεχωριστά. Μπορείτε να μας αναγνώσετε το τμήμα επί του οποίου θα ψηφίσουμε για αυτό το θέμα, σε αυτό το τμήμα. Γιατί δεν λέει στον πίνακα ψηφοφορία επί τίνο τμήματο θα ψηφίζαμε ξεχωριστά. Θα έπρεπε να είναι στον πίνακα ψηφοφορία. Ναι, αλλά δεν το λέει, λέει ο μιλητή. Λοιπόν, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει μια ρήτρα ασφάλισης ε, όπου ε, θα ε, συμπεριλαμβάνεται η εντατική πτυχή ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης για την αντιμετώπιση της διαρροής του άνθρακα και των πρώτων υλών και της χαλιβουργίας με αντίστοιχα μέτρα για την διατήρηση των δασμολογίων, τελωνιακών δασμολογίων και ποσοστώσεων όσον αφορά μια καθορισμένη μεταβατική περίοδο μετά την έναρξη σε ισχύ της TTIP με μια υποχρεωτική ρήτρα αναθεώρησης, mandatory review clause. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με αυτό το κείμενο το οποίο είναι υποψήφιση, ήτρε 6, δεύτερο τμήμα αυτής, υπέρ Παρακαλώ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την Ήτρε 6, δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Πάμε στην Ήτρε 15, υπέρ. Κατά απόχες εγκρίθηκε ήτρε 16 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε και πάμε στην ΙΜΚΟ Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΙΜΚΟ ΑΕ, σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε περνάμε στην άγκρη αιτιολογική σκέψη α υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε άγκρη Αιτιολογική σκέψη Γ υπέρ Σ υπέρ κατά θα ελέγξουμε άγκρι Σ άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε και συνεχίζουμε και πάμε στην άγρι F υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και πάμε στο Ι e, υπέρ στο I δηλαδή υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε άγρι M υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε άγρι Air. Ε, σωστό, αν το βλέπω καλά. L λοιπόν, μάλιστα. Άγκρι L. Σωστό. Καταπίπτει λέει εδώ, αν εγκριθεί η άλλη. Λοιπόν, πολύ καλά. Εντάξει, να ψηφίσουμε το L, σωστό, διότι η τροπολογία 332 δεν ψηφίστηκε. Άρα λοιπόν εκκρεμεί το Άγκρι l υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε Άγκρι ΕΛ. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 18, εγκρίθηκε όμως αυτή και περνάμε στην Άγκρι R. Άγκρι R, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίφθηκε. Περνάμε στην άγκρη γιου. Αλλά νομίζω καταπίπτει αυτή. Επειδή είχαμε μια αντίστοιχη τροπολογία της ΕΝΒΗ που εγκρίθηκε. Την ΕΝΒΗ 13 δηλαδή που εγκρίναμε. Μάλιστα. Άρα καταπίπτει αυτό. Περνάμε στη συνέχεια στην Επιτροπή Πολιτισμού. Κουλτ. Καταρχήν πρώτα έχουμε την αιτιολογική σκέψη F, κουλτ, υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Κουλτ Ή στη συνέχεια. Υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε. Κουλτ Ή. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. Εγκρίνεται. Κουλτ F. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ας ελέγξουμε. Άρχεται. Κουλτ πρώτο τμήμα του F. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Κουλτ F. Δεύτερο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κουλτ G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας, ας ελέγξουμε. Κουλτ G άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Κουλτ H υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε Τζούρι Τζούρι C Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται Τζούρι N χινιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τζούρι Q Α Καταπίπτει όχι Α ναι Α καταπίπτει ωραία Ωραία, ωραία, πολύ ωραία Λοιπόν Τώρα έχουμε λίμπε τροπολογίες Λίμπε, ε, αιτιολογική αναφορά 3. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος, όχι έλεγχος. Ας ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Λίμπε, αιτιολογική σκέψη α, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε σε τσι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα τι γίνεται με το λίμπε α να δούμε αν ισχύει ακόμη τότε να ψηφίσουμε το λίμπε α λίμπε α υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα έχουμε εγκρίνει την 617 ε, νομίζω όχι ωραία όχι οπότε ψηφίζουμε το λίμπε σε υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα αύκο λογική σκέψη α υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αύκο ε6 ή 6. Ποιοι υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Αύκο ή 8 λατινικό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε Πετή. Περνάμε στην Πέτη. Με τη λογική αναφορά 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πέτη αναφορά 4. Υπέρ. Κατά. Mm. Αποχές. Να ελέγξουμε. Αναφορά 4. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Αναφορά 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αναφορά 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σκέψη G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε την 5 14. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτω. Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο τμήμα. Τελευταίος κατάλογος προφοριών. Λοιπόν, είναι ιδεολογικές σκέψεις αναφορές. Συμβαστική 3. Ποιος την ψηφίζει. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Πρώτα έχουμε την 34. Προηγείται. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται για την τροπολογία 50 η ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οκ να ελέγξουμε την 60 άρχεται λήξη εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά Λοιπόν, ξαναρχίζω. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, κα, ε, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά Τροπολογία 78. Λέγεται ότι έχει αποσυρθεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ δεν την έχω αποσύρει. Αναφέρομαι εδώ πέρα σε ρυθμιστικέ δαπάνε και στο ρυθμιστικό κόστο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να ψηφιστεί. Yeah. Γνώμη δική μου όμω τροπολογία έχει αποσυρθεί και ήταν και αυτή μια πολύ σημαντική τροπολογία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα κρατήσουμε αυτή την τροπολογία. Αν λέω ότι έχει αποσυρθεί, έχει αποσυρθεί. Παρακαλώ πολύ ηρεμία. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει προφορική τροπολογία ανα πάσα στιγμή. Συνεπώς, αν ο κύριος Αλέζα θέλει να υποβάλει την τροπολογία αυτή ως προφορική, μπορεί να το κάνει αυτό, εφόσον δεν υπάρχει ένσταση τουλάχιστον από τρεις ευρωβουλευτές. Φαντάζομαι λοιπόν θα υποβάλει τροπολογίες προφορική και επομένω ρωτάω αυτή τη στιγμή την Επιτροπή μας αν υπάρχει κάποιος που αντιτίθεται σε αυτή την προφορική τροπολογία. Λοιπόν, δεν βλέπω να αντιτίθεται κανεί Να ψηφίσουμε το 78. Ως προφορική τροπολογία του κύριου βαλέσα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε. Την 93. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά. Παρακαλώ άλλη μια φορά ποιοι είναι κατά παρακαλώ τις 102. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ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 κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά λοιπόν επαναλαμβάνω συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 κατά αποχές εγκρίνεται τώρα περνάμε στην 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 175 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οπότε συμβαστική 10β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.27 υπέρ κατά να την ελέγξουμε είναι ταυτόσιμη με τη 2.29 ψηφίζουμε και τις δύο λοιπόν άρχεται πέρας εγκρίνεται. Οπότε περνάμε τώρα στην 28 ε, υπέρ δεν ισχύει πλέον 28; 23. Ποιοι είναι υπέρ του 23. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.31 υπέρ κατά να την ελέγξουμε 2.31 άρχεται πέρας απορρίπτεται 2.32 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα Καταπίπτει. Να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα της 2.32. Ωραία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε Ποιο είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος τώρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. Να ελέγξουμε και αυτό. Ωραία. Δεύτερο τμήμα τη 2.32. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Όχι, όχι, δεν είναι η συνήθις διαδικασία, δεν είναι η συνήθις ψηφοφορία. Είναι κατά τμήματα και για την κατατμήματα ψηφοφορία σε περίπτωση ισοψηφία εγκρίνεται. Ναι, υπήρξε κάποια σύγχυση, λέτε. Λοιπόν, και πάλι, δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 2.32. είναι αν θα πούμε με ποιον θα συζητήσουμε και ποιος είναι αρμόδιος. Και εδώ οι λέξεις Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνεται να διαγραφούν. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας, δηλαδή να διαγραφεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αν θέλετε να μείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αν θέλετε να φύγουν πρέπει να ψηφίσετε κατά. Ποιοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διατηρηθεί σε αυτήν την ε, διάταξη. Και κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όσοι θέλουν να διατηρηθεί πρέπει να ψηφίσουν συν και όσοι θέλουν να απαλληφθεί πρέπει να ψηφίσουν μείον. Και πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στη 2.33. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.35 υπέρ να ελέγξουμε το 2.34 άρχεται πέρα και απορρίφθηκε 235 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε σκεπτικό 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 2 υπέρ κατά ελέγχουμε ψηφίζουμε το, την αιτιολογική σκέψη το αιτιολογικό 2 η, άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 3 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την τροπολογία 3 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έτσι εγκρίθηκε σωστά έτσι θα έλεγα και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 15 υπέρ κατά εγκρίθηκε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 18 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 19 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 20 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 22 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 23, 24 ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 25 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27, 28, 29 είναι ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά έλεγχος ψηφίζουμε 27, 28, 29 ηλεκτρονικά άρχεται πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα εγκρίθηκαν. Χωρίς μικρόφωνο η παρέμβαση. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά αυτή τη φορά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 28 ψήφοι υπέρ 13 εναντίον εγκρίθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι ολοκληρώνουμε, κλείνει η συνεδρίασή μας για απόψε. Ευχαριστώ, γεια σας.